Αγαπητοί συνάδελφοι, αν καθυστερώ εδώ, είναι γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα με την έκθεση COX και περιμένουμε το συντονιστή από το ΕΛΚ να μας διευκρινίσει κατά πόσο ο εισηγητής θέλει να προχωρήσουμε με την έκθεση αυτή σε αυτή τη συνάντηση ή όχι. Γι' αυτό καθυστερούμε λίγο πριν ξεκινήσουμε με την εξέταση της ημερήσιας διάταξης. Επ' να καλωσορίσω ε, από, το, από την εκλογική περιφέρεια του κύριου Βαντάλεν, εδώ πίσω, καμιά εικοσαριά τομα είναι. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι συνήθως δεν έχουμε τόσο μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων. Συνήθως έχουμε πολύ μικρότερη. Τόσο το καλύτερο βέβαια που έχουμε τόσο μεγάλη αίθουσα. Συνήθω στριμωγνόμαστε ούτε αρκετέ θέσει υπάρχουν, αλλά μια που σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη αίθουσα, για σας τόσο το καλύτερο. Καλώς ήρθατε λοιπόν και χαίρομαι που σας έχουμε μαζί μας. Ωραία λοιπόν, σταματάμε για λίγο, περιμένουμε το Μάτιος να έρθει για να μας δώσει τις προφορίες περιμένουμε. herr präsident! Äh, hang on. can i formally i've not started yet i've been waiting for you so can i just formally uh, open the. περιμένω. λοιπόν καταρχήν αρχίζει η μερίσια διάταξη και τώρα έχετε διαδικαστικό σας δίνω το λόγο. ευχαριστώ πρόεδρε. ο συνάδελφος κοκ είναι στη Φραγκφούρτη ακόμα λόγω μέτρων ασφάλειας δεν θα μπορέσει να φτάσει εδώ πριν τις 6 το απόγευμα. Ξέρω όμως ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν ερωτήσεις για την εκθεσή του, για τον κατάλογο ψηφοφορίας κλπ. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίασή μας την εξέταση και την έγκριση της έκθεσης αυτής. Το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχουν ερωτηματικά ακόμα ανάμεσα στους συναδέλφους για αυτή. Αυτά έχω να πω. Ωραία. Ε, να δούμε αν κατάλαβα. Προτείνεται να βγει από την εμερήσια διάταξη η έκθεση ΚΟΚ για αυτή τη φορά. Και την εξέταση των τροπολογιών και την έγκριση. Αυτό προτείνεται και να το αφήσουμε για την επόμενη συνεδρία. Ωραία, αυτή είναι η πρόταση λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Έχει κανείς αντίρρηση από αυτού ή το δεχόμαστε. Ωραία, άρα βγαίνει από την ημερήσια διάταξη και θα μπει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασής μας. Και για όσους από εσά ήρθατε γι' αυτό, ειδικά το θέμα σήμερα, ζητώ συγγνώμη. Δεν εξαρτάται από μένα. Η, η γραμματεία πρέπει να φροντίσει να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για αύριο για τις ψηφοφορίες. Να ξέρουμε τι ώρα θα ψηφίσουμε το καθένα. Να ενημερώσουμε και την Επιτροπή, ε. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ξέρει. Καλώς. Με την αλλαγή αυτή. Α, η κυρία Μάισνερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Θέλω να καταλάβω καλά. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει τώρα η μερίσια διάταξη, αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή κάτι που προβλέπετε για αύριο το απόγευμα να πάει για αύριο το πρωί. Θέλω να το ξέρω αυτό. Θα αλλάξει και σε άλλα πράγματα η μερίσια διάταξη, απλώ αφαιρείται αυτό το σημείο. Είναι δύσκολο, λέει ο πρόεδρο, να το πω. Δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα γιατί περιμένουμε και ανθρώπου από την Κομισιόν. Ε? Οπότε εγώ θα έλεγα να τελειώσουμε νωρίτερα στις 24 και να συνεχίσουμε κανονικά στις 25 όπως έχουμε προβλέψει. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου, δεν ακούστηκε. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Εγκρίνεται με την αλλαγή αυτή το σχέδιο μερίσια διάταξη και πάλι ζητάω συγγνώμη για όσο από εσά ήρθατε για το συγκεκριμένο αυτό σημείο που αναβάλαμε. Περνάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών τη προηγούμενη συνεδρίασή μα. Συμφωνείτε. Εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ που έχει να κάνει με την ε, οδική ασφάλεια και τις παραβάσεις. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Έχεις το λόγο, Ινές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον που έδειξαν στην έκθεσή μου. Έχουν υποβάλει διάφορες τροπολογίες προκειμένου να τις ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Θα έχετε δει ότι πολλές από τις τροπολογίες δεν τις έχω λάβει υπόψη μου. Δεν τις έχω συμπεριλάβει. Και γιατί, γιατί είναι μια έκθεση αυτή για την οποία είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Διαπραγματευόμαστε με την Προεδρία, με την Κομισιόν, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Οπότε, ακριβώς επειδή θα πετύχουμε κάποιες συμφωνίες, δεν μπόρεσα να δεχτώ και όλες τις τροπολογίες που επέβαλαν οι συνάδελφοι. Προσπαθήσαμε δηλαδή να μην προσθέσουμε νέα στοιχεία. Γιατί σε άλλα πλαίσια μέσα μπορούμε να εξετάσουμε τα θέματα που θίγουν οι συνάδελφοι τώρα. Συζητάμε και την έκθεση ΚΟΧ, μην ε, ξεχνάτε. Οπότε κάποιες που είναι για την Ευρωπαϊκή Οδική Ασφάλεια, οπότε κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί πιστεύω ότι ταιριάζουν πολύ καλύτερα σε μια έκθεση πρωτοβουλίας όπως είναι αυτή του κυρίου Κόχ που κάνει συστάσεις που θέλει να συμπεριληφθούν και άλλες παραβάσεις, ε, προτείνει κυρώσεις και γενικά κάνει προτάσεις για την όλη διαδικασία ε, ανταλλαγής πληροφοριών. Ενώ εμείς για τη δικιά μου την έκθεση προχωράμε καλά με την Προεδρία. Οπότε αν προσθέσουμε τροπολογίες που, είναι, που πρόκειται να προσθεθούν στα ήδη δύσκολα θέματα που ε, διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο θα έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο οι διαπραγματεύσεις αυτές. Ζητώ συγγνώμη, γιατί πριν από δύο εβδομάδες ήδη πρόκειτο να παρουσιάσω τι δυνατότητες υπάρχουν για συμβαστικές τροπολογίες. Για παράδειγμα για τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τις κατεξουσιοδότηση πράξη της κυρίας Τικάου ή για την προστασία δεδομένων του κύριου Μπάχ, Σάφισαρ, Ρικέτ κλπ. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα. Γιατί είχαμε τη, στη συζήτηση με την, για την Ευρωβινιέτα να αναβληθούν τα θέματα αυτά από την Κορεπέρ και η Προεδρία δεν μπορούσε να μας πει κατά πόσο είχε εντολή για να συνεχίσουμε ή όχι. Σήμερα συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω στο κείμενο. Οπότε μπορώ να σας πω ότι για την προστασία δεδομένων για τις κατεξουσιοδότηση πράξης έχουμε προχωρήσει πολύ. Μάλιστα το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να θέσει την αναγκαιότητα να υπάρξουν μέχρι και ενιακριτήρια, κριτήρια, εναρμόνιση. Αλλά σήμερα το πρωί, εν πάση περιπτώσει, στον τριμερή διάλογο δεν μπορέσαμε να υποβάλουμε συμβιβαστικές τροπολογίες όπως θέλουμε για να πάμε με αυτές την Ολομέλεια. Οπότε για άλλη μια φορά ζητώ κατανόηση από τους συναδέρφους. Πολύ θα ήθελα στο κατάλογο ψηφοφοριών να είχα συμπεριλάβει και συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά έτσι όπως έχει η κατάσταση, που δηλαδή συναντήσαμε περισσότερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις, δεν το καταφέραμε. Όμως προτείνω να προτείνετε τις ε, τροπολογίες σας στην έκθεση ΚΟΧ. Εκεί νομίζω ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Αυτά, Πρόεδρε. Δεν έχω τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα περιμένω ό,τι ερωτήσει έχουν οι συνάδελφοι με στη διάθεσή τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Πάχ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ευχαριστήσω και θα συγχαρώ την κυρία Αιάλα Σέντερ για την πολλή δουλειά που έκανε καθώς και για τις συμβαστικές της τροπολογίες τις οποίες υποστηρίζουμε. Το θέμα είναι δύσκολο και ήδη μας απασχολεί εδώ και καιρό. Ασφαλώς δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί η μεγάλη αντίσταση των χωρών μελών. Γι' αυτό και την συγχαίρω. Είναι κρίμα που δεν μπόρεσε να συνεχίσει να εργάζεται στη γνωστή νομική βάση της ασφάλειας στις χερσαίες μεταφορές και χρειάστηκε να μεταφέρει την βάση στην αστυνομική συνεργασία. Δηλαδή τις ε, συνθήκες πριμ που λαμβάνει εν τέλει το θέμα διαφορετική τροπή από αυτήν που επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όντας πλέον φιλόδοξο ήθελε ανάληψη πρωτοβουλειών που να υπερβαίνουν τα όρια αυτών των συμβάσεων. Είναι λοιπόν κρίμα που λόγω της νομικής βάσης δεν δεσμεύονται τρεις χώρες από την απόφαση αυτή. Η κυρία Γιάλα Σέντερ είπε ότι η προστασία των δεδομένων είναι σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε σταθεροί και θα πρέπει να είναι αυστηροί και ικανοί στο διέπουν αυτή την προσωρινή τήρηση των δεδομένων. Επίσης σημαντικές ήταν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ουγγρική Προεδρία επίσης στην αξία συγχαρητηρίων διότι εξ αρχής ήταν δύσκολο το έργο της νομίζω όμως ότι οι τελευταίες συναντήσεις του τριμερούς διαλόγου επέτρεψαν να ευρεθούν λύσεις σε πολλά θέματα και να υπάρξει συμφωνία. Μένει τώρα αυτή η υποχρέωση κοινοποίησεως, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ δεν ικανοποιήθηκε πλήρως. Πρέπει να συζητήσουμε ακόμη δηλαδή, γιατί είναι σημαντική αυτή η υποχρέωση κοινοποίησεως από πλευρά της χώρας μέλους, δηλαδή τι μορφή θα πάρει και πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πάντως, συνολικά θεωρώ ότι η εργασία ήταν σημαντική, οι συμβαστικές λύσεις που τελικά προτείνονται είναι σημαντικές και ενδιαφέρουσες και νομίζω ότι μπορούμε στο σύνολο να είμαστε ικανοποιημένοι με την εργασία αυτή. Ευχαριστώ. Κύριε Σάβησα, για τους εξονόματος των φιλελευθέρων. Εγώ Ήδη, κύριε Πρόεδρε, έχω εκφράσει την απογοήτευσή μου για την παρούσα οδηγία. Παρ' όλα αυτά θα ευχαριστήσω την εισηγήτρια, η οποία επετέλεσε θαυμάσιο έργο, έδειξε πνεύμα συνεργασίας με τους σκιώδεις εισηγητές και εν τέλει καταλήξαμε στο σημείο που μπορούμε αύριο να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Θα έρθω τώρα ε, στην ουσία. Μιλούμε για κυρώσεις, αλλά οι κυρώσεις δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία. Νομίζω ότι για την τροχαία ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό να υφίσταται κυρώσεις όσοι διαπράττουν αδικήματα. Ελπίζω ότι βλέπουμε απλώς την απαρχή μια προσπάθειας και ότι θα μπορέσουμε εν τέλει να καταλήξουμε στους στόχους που έχουμε βάλει από την αρχή. Και όταν θα έρθουμε στις τροπολογίες, προστασία δεδομένων δηλαδή, καθώς και η κοινοποίηση, και παρόλο που το Συμβούλιο λέει ότι η προστασία δεδομένων καλύπτεται από διάφορες οδηγίες και άλλες αποφάσεις, εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι επαρκές. Θα πρέπει οι οδηγίες να λένε καθαρά ποιος έχει το δικαίωμα να ζητεί τα δεδομένα και για ποιο συγκεκριμένο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν αυτά. Θα πρέπει να, να, να, να αναφέρονται σε πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, αλλά επίσης και σχετικά με τις υποχρεώσεις των προσώπων που ενέχονται. Ο κύριος Μπαχ και εγώ έχουμε καταθέσει τροπολογίες κυρίως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και εγώ μάλιστα έχω καταθέσει και τρεις τροπολογίες για το παράρτημα. Οι τροπολογίες 70 και 71 εξετάζουν την επιστολή κοινοποίηση και η τροπολογία 72 αναφέρεται στο δεύτερο παράρτημα, παράγραφος 8 Το θέμα της έρευνας θα πρέπει να αναφέρεται μοναχά στο κείμενο του Συμβουλίου. Όλες οι χώρες μέλη δεν απαραίτητο να διαθέτουν ε, πληροφορίες για ολόκληρη την υπόθεση, διότι μόνο η χώρα εκείνη στην επικράτεια της οποίας τελέστηκε το αδίκημα θα πρέπει να έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να ε, συλλέγει τα δεδομένα. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια πραγματικά κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια. Το Συμβούλιο Υπουργών δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια. Το Συμβούλιο Υπουργών το μόνο που θέλει είναι κάθε προσπάθεια βελτίωσης της νομοθεσίας που ξεκινά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την καταδικάζει σε αποτυχία. Μόνο αυτό ενδιαφέρει το Συμβούλιο. Και ειδού το παράδειγμα. Είναι η παρούσα υπόθεση. Τι μένει τώρα, βελτίωση της ε, διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών και η υπόθεση της καταχώρησης σε Μητρό. Πράγματα δηλαδή τα οποία απέχουν πολύ από αυτά που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η τροχή ασφάλεια. Έχετε δίκιο κυρία Τόμας όταν λέτε ότι ένα από τα κύρια θέματα είναι το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Οι διατυπώσεις που έχουμε τώρα μπροστά μας επιτρέπουν σε μια ε, χώρα μέλος να διατηρεί τα δεδομένα αυτά για 13 χρόνια. Διότι δεν υπάρχουν de facto καθορισμένες, καθορισμένα μάλλον όρια. Άρα κάθε υπόθεση θα καταλήγει ενώπιον των δικαστηρίων. Μα δεν πρέπει εδώ να νομοθετούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλούνται κατόπιν τα δικαστήρια να ε, ξεκαθαρίζουν την ομολογία αυτή. Αυτά που κάνει λοιπόν το Συμβούλιο έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα και γι' αυτά διόλου δεν βαρύνεται η κυρία Αγιάλα Σέντερ η οποία έκανε πολύ καλή δουλειά η οποία όμως απέτυχε λόγω της αδράνειας του Συμβουλίου. Επιτύχαμε μόνο μία μικρή βελτίωση. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να διατυπωθεί με τέτοια ακρίβεια η προστασία των δεδομένων, ώστε να μην μπορεί να γίνει καμιά κατάχρηση από πλευρά χώρων μελών. Διότι περί αυτού εν τέλει πρόκειται. Ότι δηλαδή τα δεδομένα αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ιονδήποτε σκοπό, παρά μόνο για τον σκοπό για τον οποίο διατίθεται, για τον οποίο συλλέγονται. Από τις πολλές διατυπώσεις μας τελικώς μένουν μονάχα δύο παράγραφοι, οι οποίες μάλιστα είναι και αντιφατικές μεταξύ τους και όχι εκτελεστές, διότι εν τέλει θα καταλήξουμε τα πράγματα να παραμείνουν όπως είναι. Και αυτό μάλιστα τέτοια πράγματα δηλαδή δεν σημειώνονται μονάχα σε θέματα μεταφορών. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να παράγει νομοθεσία η οποία είναι απαραίτητο να διαλευκένεται στα δικαστήρια. Πρόκειται δηλαδή καθαρά για παράδειγμα του πως δεν θα έπρεπε να γίνονται τα πράγματα αυτά. Το άλλο είναι βεβαίως η περίφημη ευρωβινιέτα. Εδώ όμως πρόκειται για θέματα τα οποία δεν μπορούν να περιπληθούν τον μανδύα των διμερών συμφωνιών. Και είναι πραγματικά διανοητική παινία του Συμβουλίου. και ούτε καν ευθύνεται μοναχά η Προεδρία του Συμβουλίου. Είναι η γενική πολιτική του Συμβουλίου που λέει «Α, ναι, ωραία, έχει αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα τώρα το Κοινοβούλιο στη βάση της συνθήκης της Λισαβόνας, θα το αποδείξουμε και εμείς, το Συμβούλιο δηλαδή, ότι αυτά είναι μονάχα στα χαρτιά, εμείς είμαστε τα αφεντικά και θα καταστρέψουμε κάθε πρωτοβουλία που προέρχεται από τα δικαιώματα αυτά». Πρόκειται δηλαδή καθαρά για τυπικά παραδείγματα τέτοιας αδράνειας. Ο κύριος Βαντάλια από Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια. Έχουμε την άποψη ότι η συγκίτρια έκανε ό,τι πέρναγε από το χέρι της για να καταφέρει να φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Μπορώ να καταλάβω αυτά που λέει η συγγήτρια, ότι της ήταν δύσκολο να προχωρήσει με τις τροπολογίες μας. Ήταν... Είναι πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, οπότε λέω ότι θα γινόντουσαν ακόμα πιο δύσκολες αν έβαζες αυτές και τις καινούργιες τροπολογίες. Όμως θέλω να ζητήσω να προσέξετε την τροπολογία Μπαχ και δικιά μου. Μέχρι την 51 που εμείς μιλάμε για ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται στην εθνική νομοθεσία. Και γιατί, γιατί ορισμένες χώρες δουλεύουν με διαφορετικούς τρόπους όσον αφορά την ε, δίωξη. Αλλού γίνεται μια συνεννόηση, αλλού ζητάνε χρήματα, βάζουν πρόστιμα, αλλού είναι ποινικέ οι διαδικασίες. Οπότε με τον συνάδελφο Μπαχ έχουμε πει ότι θέλουμε ένα σύστημα συγκεκριμένο για όλες τις χώρες. Δυστυχώς η συγκήτρια δεν το στηρίζει αυτό. Ίσως θα μπορούσε να μας απαντήσει πάνω σε αυτό. Πάντως θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους να προσέξουν όλους ιδιαίτερος τις τροπολογίες αυτές 50 και 51. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρικέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, την Ινέση για τη δουλειά της. Ξέρω και εγώ ότι είναι δύσκολη η δουλειά της. Οι τροπολογίες που πρότεινα εγώ, προφανώς το Συμβούλιο δεν τις έλαβε υπόψη του καθόλου. Κι όμως πρόκειται για ένα βασικό δικαίωμα. δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζουμε μια ποινική ε, καταδίκη εναντίον κάποιου βασιζόμενη στο ε, όχημα, στα στοιχεία του οχήματο και μόνο. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στη φυλακή τον ιδιοκτήτη του οχήματο για ένα ποινικό αδίκημα που ενδεχομένω δεν έκανε ο ίδιο. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι όντω έχουμε ενημερώσει σχετικά αυτόν που διέπραξε την παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν έκανα και την πρότασή μου. Τελικά έχει καταλήξει στα σκουπίδια. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα κάποιος να υποστηρίξει ότι όντως δεν έχει πάρει ε, την ε, ειδοποίηση για την παράβαση που έκανε. Είναι ένα σύστημα δηλαδή που δεν αρκεί. Ε, χρειάζεται ένα συστημένο. Με την πρόταση έτσι όπως έχει τώρα υπάρχουν τρεις αρχές. Πρώτον, ότι καταδικάσουμε κάποιον βάσει το οχήματο ή όχι. Τρίτον, ότι η ποινική διαδικασία δεν ακολουθείται όπω πρέπει. Και τρίτον, ε, παραβιάζεται το απόρριτο. Είναι τρει αρχέ που παραβιάζονται με την πρόταση αυτή. Και εμένα με εκπλήσει άσε που δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί έχει να κάνει με παράβαση και του εθνικού δικαίου και του ευρωπαϊκού. Οι χώρες που αντιτίθεται στην εφαρμογή διασυνοριακών κυρώσεων τελικά θα κερδίσουν, γιατί η οδηγία αυτή δεν θα μπορέσει ποτέ να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Ευχαριστώ. κυρία Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ενώ θυμίζω την γνωστή θέση της Κομισιόν Οικονομική Βάση θα ήθελα να σας πω ότι καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το σημαντικό ε, φάκελο για την οδική ασφάλεια και την ε, σχετική πολιτική της Ένωσης. Συμφωνώ ότι έχει σημειωθεί θετική πρόοδος και η Κομισιόν είναι πολύ αισιόδοξη ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση τον Ιούλιο. Έχει γίνει πολλή δουλειά τους τελευταίους μήνες και θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος της Κομισιόν την εισηγήτρια καθώς και την Ουγγρική Προεδρία διότι η προσέγγιση της είναι πολύ επικοδομητική και έχει οδηγήσει ήδη σε σημαντικές υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, κυρίως όσον αφορά τη ρήτρα αναθεώρησης και τη ρήτρα περί προστασίας δεδομένων. Ούτως ή άλλως θα ήθελα να στραφώ σε κάποιες τροπολογίες που αναφέρατε εδώ ήδη. Εμεί καλωσορίζουμε την ενδυνάμωση της υποχρέωση των κρατών μελών να, αναφέ, να κάνουν αναφορά, τροπολογία 18, για την 17, για την επιστολή την ενημερωτική. Ξέρουμε πω είναι δύσκολο να συνδυάσει ε, δύο απόψεις ε, διαφορετικές νομοθετικές, αλλά είμαστε θετικοί όσον αφορά τη συμβαστική λύση που κατατέθηκε σήμερα. Επίσης θα σας δώσουμε τα αποτελέσματα στον επόμενο τριμερή διάλογο που θα γίνει στις 7 Ιουνίου. Επίσης πιστεύουμε ότι η υποστήριξη για πιο ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης που όπως προτείνεται στην τροπολογία 25 ε, και αναφέρεται στις κατευθύντηρες γραμμές και την εναρμόνιση των ε, ε, κατευθυντηρίων γραμμών προβλέπει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της ε, Κομισιόν. Και εδώ φυσικά έχουμε υπόψη μας τη σημασία αυτής της ζήτητας αναθεώρησης ε, για το Κοινοβούλιο και είμαστε σύμφωνοι με τη λύση που έχει βρεθεί. Ε, τώρα, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, πιστεύουμε ότι ναι, πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά τα περισσότερα, οι περισσότερες από τι του Ευρωκοινοβουλίου έχουν ήδη ληφθεί υπόψη Άρα μια τεχνική λύση για τις λεπτομέρειες θα βρεθεί. Η Κομισιόν επίσης σημειώνει την διάταξη για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση ενώ υπάρχει κοινή συνεννόηση για τις ε, κατεξοδόσεις της πράξης ε, παρέχουν μια επιλογή, παρέχει μια επιλογή για κοινή λύση. Και να τονίσω η τροπολογία 52 που αφορά την προστασία των στοιχείων. Ε, να σας πω ότι η Κομισιόν συμφωνεί για το πρώτο τμήμα, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσει ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί για να εποφύγουμε οποιαδήποτε μπλοκές σε μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις και οι τροπολογίες 50 και 52 πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν μια κάποια νομική αβεβαιότητα να, πρέπει να ξαναδιατυπωθούν δηλαδή και για τη 49 νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να αποδυναμώσει τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτή είναι μια αρχική θέση την οποία μπορούμε να σας δώσουμε και μετά από το σημερινό τριμερή διάλογο όπως ήδη τονίσαμε η Κομισιόν είναι πολύ αισιόδοξη και θετική ότι δηλαδή στον επόμενο τριμερή διάλογο θα βρεθεί επιτυχής και θετική λύση για την οδική ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσπαθεί να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουμε στον τριμερή διάλογο. Θέλω να πω στον κύριο Μπόχ ότι όντως επειδή χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα το Συμβούλιο μπλόκαρε τα πράγματα θελήσαμε να προσπαθήσουμε με μια άλλη νομική βάση να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και η Προεδρία, η Βέλγικη Προεδρία βοήθησε πολύ διότι μπήκαμε από άλλη οπτική γωνία να εξετάσουμε ένα θέμα πολύ βασικό. Επίσης, κάτι άλλο που καταφέραμε στον τριμερή διάλογο είναι, όπως έλεγε η κυρία Γέγερ πολύ σωστά, να έχουμε μία ρήτρα αναθεώρησης για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη νομική βάση μεταφορές. Οπότε στο μέλλον οι νέες προτάσεις που θα χρειαστούν θα γίνουν με τη νομική βάση μεταφορές. Έτσι το Συμβούλιο δέχεται να συνεχίσουμε. Τρεις χώρες, η Δανία για παράδειγμα δεν ήθελε να συμπεριληφθεί, αλλά το Ενωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία είπαν πως ναι και κυρίως και γι' αυτό και ευχαριστώ και την Ουγγρική Προεδρία γιατί στο παράρτημα 1, το τεχνικό παράρτημα επίσης που τίθεται το θέμα του ποινικού συστήματος και της ανταλλαγής πληροφοριών και μιλάμε για προσαρμογή της ανταλλαγής δεδομένων όταν πρόκειται για παραβιάσεις του οδικού κώδικα οι τρεις χώρες ε, που αρχικά είπαν ότι μένουν απ' έξω θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα και εφόσον τελικά κάποια στιγμή το θελήσουν. Γιατί εμεί δεν θέλουμε να σταθούμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο ε, βάσει το οποίο δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι αυτοί που στο μέλλον θα θελήσουν να το χρησιμοποιήσουν θα μπορούν. Για την προστασία δεδομένων. Όντω είναι ένα από τα σημεία στα οποία έχουμε κολλήσει κάπως στο Συμβούλιο. Υπάρχει γενική ρήτρα για την προστασία δεδομένων, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει ειδικότερα να δούμε τη νομική βάση της αστυνομικής συνεργασίας που απαιτεί μεγαλύτερη προστασία δεδομένων γιατί πρόκειται για εγκλήματα ή για την τρομοκρατία. Λοιπόν, πρέπει να προσαρμόσουμε τα πράγματα στο δικό μας θέμα που είναι η οδική ασφάλεια. Και γι' αυτό χρειάζεται κάτι να γίνει. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο θα δεχτεί, ελπίζουμε να το δεχτεί, το έλεγα και στον Λίχτεμπεργκερ, στην κυρία Λίχτεμπεργκερ, ότι θα δεχτεί προθεσμίες για να μπορέσει να γίνει ανταλλαγή δεδομένων με αρκετή προστασία. Έρχομαι τώρα στο παράρτημα που θέλει η κυρία Σαφιζάρη να τροποποιηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων. Πρέπει να τη πω ότι είναι ένα παράρτημα που ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω ότι και με όλα τα άλλα τα στοιχεία για την προστασία δεδομένων θα μπορέσουμε να ελέγξουμε καλά οποιαδήποτε περίπτωση κατάχρησης. Δεν χρειάζεται να μπει στο κύριο σώμα. Υπάρχει αρκετή ασφάλεια ώστε να αποφύγουμε κατάχρηση των στοιχείων. Κύριε Βαντάλεν, σας ευχαριστώ για την τροπολογία σας που είναι όπως και εκείνη του κυρίου Μπαχ. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση της, του εντοπισμού του ιδιοκτήτη του οχήματος, αυτή είναι η μόνη βεβαιότητα που έχουμε. Δηλαδή υπάρχει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ε, έχει το πιστοποιητικό ταξινόμησης του οχήματός του βάσει του αριθμού κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Το πρόβλημα είναι για τις χώρες μέλη που απαιτούν να δεχτούμε ότι ο ιδιοκτήτης είναι και ο οδηγός τη στιγμή της παράβασης. Εκείνη που χρειάζεται μια κάποια διευκρίνηση. Πάντως γι' αυτό που απασχολεί τον κύριο Φαντάλη, νομίζω ότι καλύπτεται. Τέλος να πω και στον κύριο Ρίκε ότι το να καταδικάσουμε κάποιον επειδή έχουμε εντοπίσει το αυτοκίνητό του Κοιτάξτε, εμείς χρησιμοποιούμε την νομική βάση της αστυνομικής συνεργασίας και ένα σύστημα που ακριβώς απαιτεί όλες τις εγγυήσει. Όλο αυτό το σύστημα ασφάλειας και προστασίας ώστε ο εντοπισμός να γίνεται έτσι ώστε να υπάρχει και νομική ασφάλεια όπως στη Γαλλία είναι κάτι που μας δίνει περισσότερες εγγύσεις, όχι λιγότερες. Δεδομένου ότι τα ταχυδρομεία καλύπτονται από κάποια διοντολογία προστασίας δεδομένων. Δεν νομίζω ότι κανείς θα κάτσει και θα διαβάσει ε, το γράμμα με το οποίο φτάνει το πρόστιμο. Άλλοι τα στέλνουν συστημένα, άλλοι δεν τα στέλνουν συστημένα, εξαρτάται από χώρα σε χώρα. Εμείς λέμε εθνική νομοθεσία. Ό,τι λέει εθνική νομοθεσία, έτσι καθησυχάζουμε τα κράτη-μέλη. Αυτοί που έχουν περισσότερες εγγύσεις μπορούν να τις κρατήσουν και αυτοί που θέλουν να βελτιώσουν τις δικές τους εγγύσεις και να τις κάνουν ακόμα μεγαλύτερες μπορούν έτσι να το κάνουν. Το αν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη είναι αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο είχε προβλέψει μια πλήρη διαδικασία εξετάζοντας όλες τις δυνατότητες. Δεν συμφώνησε το Συμβούλιο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να περιμένουμε το Συμβούλιο να ε, μπορέσει να προχωρήσει. Και έχει γίνει σε έναν βαθμό. Για να καταπολεμηθεί η ατιμορρησία τα κράτη-μέλη, αν μη τι άλλο, δεν μπορούν να πούν ότι η Ευρώπη δεν τους βοήθησε, δεν τους έδωσε ένα μέσο για να μπορούν να εντοπίζουν τους υπεύθυνου. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να προχωρήσουν και σε δίωξή του. Τους επιτρέπουμε όμως, τους δίνουμε τα μέσα που χρειάζονται για να το κάνουν. Είναι ένα πρώτο βήμα. Στα πέντε χρόνια και το Συμβούλιο έδωσε αρκετά στοιχεία και η Επιτροπή τα χρησιμοποίησε και μπορεί να αξιολογήσει τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά αυτά τα χρόνια και από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια. Έπειτα υπάρχει και αυτή η ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης που θα μας επιτρέψει να πάμε ακόμα πιο μπροστά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Επόμενο σημείο στην ημέρηση διάταξη είναι η δική μου έκθεση. Για όσους αργήσαν έχουμε αφαιρέσει την έκθεση ΚΟΚ γιατί δεν είναι εδώ ο κύριος Κοκ. και αυτή είναι η δική μου έκθεση για τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων. Να σας θυμίσω ότι πρόκειται για μια καθαρά τεχνική φύση έκθεση. Η Κομισιόν πρότεινε μια αναδιατύπωση ώστε καταρχήν να κωδικοποιηθούν οι διάφορες πράξεις που ισχύουν για τις στατιστικές μεταφορών ε, οδικών μεταφορών και έπειτα για να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία στο να θέσουμε κάποιες νέους όρους για την κατεξουσιοδότηση πράξης. Εγώ έχω υποβάλει 13 τροπολογίες ως ε, τμήματα του σχεδίου έκθεσης και δεν υπάρχει αλλαγή όσον αφορά το περιεχόμενο. Όλες οι τροπολογίες αφορούν τις πράξεις κατεξουσιοδότηση και τις εφαρμοστικές πράξεις. Ε, και είναι σύμφωνε με τι θέσει του Κοινοβουλίου. Για κάποιε από τι τροπολογίε για τι πράξει κατεξουδότηση έχω χρησιμοποιήσει την ίδια διατύπωση όπω αυτή που συμφωνήσατε ε, εσείς και το Συμβούλιο για τις στατιστικές περί τουρισμού. Για παράδειγμα, υποχρέωση της Κομισιόν να συμβουλεύεται εμπειρογνωμόνες ε, και όχι εθνικούς εμπειρογνώμονες και έπειτα αλλάζει μέσω των ε, κατεξοδότηση πράξεων θα πρέπει να περιορίσει το οικονομικό άχθος των ε, υπόχρεων ε, υποβολή στατιστικών στοιχείων. Επίσης, στόχο έχουμε να περιορίσουμε το εύρος των αρμοδιοτήτων που αναθέτουμε στην Επιτροπή. Τα υπόλοιπα είναι απλώς προσαρμογές στις διατυπώσεις. Τώρα, όσον αφορά τις πράξεις κατά Οι νέοι κανόνε που χρησιμοποιούν η γραμματεία μπορεί να χρειαστεί να τελειοποιηθούν από τους ε, νομικούς γλωσσολόγου μα εδώ στο Κοινοβούλιο. Και εκτό από τι δικέ μου τροπολογίες υπήρξαν 14 τροπολογίες που υποβλήθηκαν στο σχέδιο έκθεσης. Το βασικό κομμάτι είναι τη κυρία Λίχτεμπεργκερ που προτείνει τροπολογίε που έχουν επίπτωση στο περιεχόμενο του κανονισμού και τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται. Η εγκυρότητα, η μάλλον τη δημοσίευση προτείνει ότι τα στοιχεία που θα πρέπει να συλλέγονται να δημοσιεύονται το αργότερο 12 μήνε μετά από το έτος και το τρίμηνο στο οποίο αναφέρονται. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό με αυτή την τροπολογία. Η κυρία Λιχτεμπέργκερ επίση προτείνει να συλλέγονται νέα σε στατιστικέ μεταβλητέ όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ τάξει ε, οχημάτων, του ταχογράφου, του ψηφιακού ταχογράφου, ε, το φορτίο και την υπερφόρτωση που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν τα οχήματα. Αυτή είναι η εντολή της πρότασης. Η διαδρομή και τα εμπορεύματα που μεταφέρονται. Εγώ συνομίλησα με την Κομισιόν για να πάρω την άποψή τους για αυτές τις τροπολογίες και η άποψή τους είναι ότι και οι προσθήκες της κυρίας Λιχτεμπεργίας δεν είναι σύμμορφες προς τις πληροφορίες που συλλέγονται με βάση αυτόν τον κανονισμό που λένε ότι στόχο έχει να στηρίξει το εμπόριο και την οικονομία της Ένωσης. Ωστόσο, εγώ δεν είμαι αντίθετο στο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερες στατιστικές και να διευρύνουμε τη συλλογή των στοιχείων σε τομείς που είναι σχετικοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά στοιχεία. Εγώ θα στηρίξω λοιπόν τις τροπολογίες της κυρίας Λιχτεμπέργκερ για τη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά το Τη κλάση των αυτοκινήτων, τον ψηφιακό ταχογράφο και πιστεύω πω επίση θα υπάρξει μια προφορική τροπολογία από την κυρία Λίχτεμπεργκερ για να αποσαφινιστεί η θέση μα σε σχέση με αυτό το σημείο. Ταυτόχρονα θα χρειαστεί να βάλω ένα πλήν σε κάποιε από τι τροπολογίε, γιατί υπάρχουν βάσιμοι λόγοι γιατί οι πληροφορίες αυτές δεν είναι σχετικές με αυτόν τον κανονισμό. Υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας. Τα βασικά στοιχεία που δίνονται από τον ίδιο τον οδηγό Άρα λοιπόν ε, το να συλλέξουμε στοιχεία για τον χρόνο ανάπαυση ή την υπερφόρτωση δεν θα λειτουργούσε εδώ. Τώρα για τα σοβαρά ατυχήματα τα στοιχεία αυτά ήδη συλλέγονται με την 704 του 93 την οδηγία του Συμβουλίου. Τέλος θα θυμίσω και την ε, τροπολογία 17 της κυρίας Τικάου και αποσύρω τη δική μου 7 που καλύπτει το ίδιο θέμα γιατί η διατύπωση της κυρίας Τικάου είναι πιο ενήμερη και αντικατοπτρίζει την ισχύουσα διατύπωση περί πράξεων κατεξουδότηση. Εν κατακλείδη λοιπόν, θα ήθελα να πω επίσης ότι η τροπολογία 15 του κυρίου Μπαλσάιτης μου φαίνεται κάπω περιττή, γιατί μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν ούτω ή άλλω να συλλέγουν στοιχεία σύμφωνα με τη διαδικασία που καταγράφεται, γιατί διαφορετικά θα παραβίαζαν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Υποστηρίζω λοιπόν την, από έσυρα την 7, υποστηρίζω λοιπόν την 17 της κυρίας θα υποστηρίξω και την τροπολογία 16 της κυρίας Λίχτεμπεργκερ και τις τροπολογίες 18 και 19. Αυτά είχα να πω για το θέμα. Ο κύριος Γκρός από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα υποστηρίξουμε σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις σας καθώς και τις τροπολογίες σας και όσον αφορά τις τροπολογίες της κυρίας Λίχτενμπέργκερ θα συμφωνήσουμε με την υπαριθμόν 18 για τις κατηγορίες εκπομπών καυσαερίων για την 19 ίσως είναι καλύτερο να γίνει μια ακριβέστερη διατύπωση που φαντάζομαι ότι θα γίνει για την 16 Καλό είναι να γίνει το έτος μετά από το έτος αναφοράς. Αλλά το ερώτημα είναι πότε θα δοθούν τα δεδομένα, έξι μήνες μετά. Θα προτιμούσα λοιπόν να γράψουμε το έτος μετά από το έτος ε, κοινοποίησης των δεδομένων. Για να υπάρχει και ένα διάστημα για να γίνει σχετική εξέταση. Κατά τα άλλα, οι πληροφορίε είναι σημαντικές, αλλά υπάρχουν και κάπου αλλού. Αυτό αφορά τις τροπολογίες 20, 21 και ενδεχομένω και 22. Και δηλαδή τα δεδομένα της Ευρωστάτ για τα ατυχήματα. θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση με τις υφιστάμενες πληροφορίες. Αυτό βέβαια να γίνει εκ παραλίλου, για να μην υπάρξει επικάλυψη εργασίας. Άρα, σε μεγάλο εύρος θα υποστηρίξουμε τις προτάσεις αυτές. Μάισνερ, κυρία Μάισνερ. Θα είμαι σύντομη έστω και αν αυτό οδηγήσει να είναι συντομότερη συνεδρίαση διότι στην λίστα ψηφοφοριών θα συμφωνήσουμε σε όλα με τον εισηγητή τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα και με πολύ παρόμοια αιτιολογία που δεν θα την επαναλάβω επομένω. Είναι λοιπόν σημαντικό που έγιναν τροπολογίες από τον εισηγητή σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που έχει να δράσει αυτόνομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσέξουμε τι θα γίνει με τις διάφορες τροπολογίες ε, της κυρίας Λίχτενμπέργκερ και εκεί συμφωνώ πάλι με τον εισηγητή διότι δεν είναι σωστό να γίνει επικάλυψη χορήγησης δεδομένων και να δούμε και από αυτά τα πράγματα που ζητούμε ποια ε, είναι τα πιο σημαντικά. Άρα Θεωρώ ότι η... είναι σωστή η έκθεση. Η γραμμή είναι σωστή και την υποστηρίζουμε. Η πορεία δηλαδή. Ευχαριστώ, Λίχτενμπεργκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που υποστηρίζουν ορισμένες από τις τροπολογίες μου. Θα σας εξηγήσω ποια για ποιο λόγο τις ε, υπέβαλα. Είχαμε αποφασίσει στην τελευταία περίοδο να ζητήσουμε σύνταξη εκθέσεω για τις ε, ώρες εργασίας και αναπαύσεως και για το εάν η πυκνότητα των ελέγχων που ζητήσαμε και ε, ως Επιτροπή δηλαδή και τελικά έγιναν δεκτές εάν όντως τηρούνται από τις χώρες μέλη. Και εδώ τέθηκε το θέμα της προθεσμίας το 2007 ή, ε, το 2007 ή 2008 ήταν αυτό, ζητήσαμε ε, ε, δεδομένα και απεδείχθη ότι μόνο τα δεδομένα μέχρι το 1999 ήταν πλήρη. Ορισμένες χώρες λοιπόν δεν κοινοποιούν δεδομένα. Και γι' αυτό μου φαίνεται ότι η ιδέα του κυρίου Γκρός, δηλαδή να λέμε ένα χρόνο μετά την παράδοση των δεδομένων, πάλι δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε, διότι κάποιες χώρες δεν θα ε, κοινοποιήσουν τα δεδομένα και αν χρειαστεί να περιμένουμε να κοινοποιήσουν τα δεδομένα όλες οι χώρες θα έχουμε καθυστέρηση ίσως και μιας δεκαετίας και τότε δεν χρειάζεται καν να κάνουμε την προσπάθεια. Δηλαδή ε, άδικος σκόπος. Εγώ λοιπόν θέλω να στο ευρωπαϊκό επίπεδο η έλεγχη αυτή των οχημάτων όπου δεν υπήρχαν δεδομένα νεότερα της πενταετίας. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει κανείς ούτε και προβλέψεις στον τομέα των χερσιών μεταφορών διότι αλλάζουν πολλά πράγματα λόγω της, ανανέωσης των, ε, της τεχνολογικής ανανέωσης των οχημάτων. Να δώσουμε λοιπόν συνολικά δεδομένα για ό,τι αφορά τις ε, μεταφορές εμπορευμάτων οδικός. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να γίνει επικάλυψη δηλαδή διπλή συλλογή των δεδομένων αυτών. Εάν πάντως έτσι το βλέπουν κάποιοι, με ενδιαφέρει να το συζητήσω. Και σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τους ταχογράφους, η αιτιολογία είναι, είχαμε συζητήσει τότε σχετικά με την εισαγωγή των ταχογράφων, τους διάφορους τύπους. Αλλά είπαμε, ας δούμε πόσα οχήματα θα πρέπει να εξοπλιστούν με ταχογράφους και είπα εν τέλει να βάλουμε ψηφιακή ταχογράφη ή ψηφιακούς ταχογράφους στο κείμενο. Επισημαίνω μόνο ότι ορισμένα δεδομένα συλλέγονται μονάχα σε επίπεδο των χωρών μελών και πάλι όχι όλων των χωρών μελών. Και γι' αυτό εν τέλει δεν έχουμε βάση για λήψη αποφάσεων σε πολλά θέματα. Θυμίζω και την συζήτηση για την Ευρωβινιέτα. Πόσα οχήματα, δηλαδή ακόμα ευρω, ευρωπροδιαγραφών 3 και 4 κυκλοφορούν ακόμη στους δρόμους. Θα ήταν βέβαια σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, διότι αλλιώ θα εγκρίνουμε κάποια ρύθμιση για την Ευρωβινιέτα, η οποία θα αφασίζεται σε κάτι το οποίο δεν υφίσταται πλέον. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι ανταποκρίνεται στο better making στην προσπάθεια να δηλαδή, βελτίωση της νομοθεσίας. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα να λαμβάνουμε, να μας κοινοποιούνται τα δεδομένα το δυνατόν εγκαιρότερα. Διότι η συνήθιση ύποπτη είναι γνωστή. οι χώρες δηλαδή οι οποίες ίσως κοινοποιούν δεδομένα με καθυστέρηση μιας δεκαετίας, ίσως και καθόλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ δεν είναι βεβαίως να εργαστούμε ως ιστορικοί του παρελθόντος, παρόλο που καμιά φορά μου φαίνεται ότι αυτό ακριβώς πάμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Σέλερ θέλετε να μιλήσετε, όχι. Καλά. Ευχαριστώ και χαίρομαι που μπορέσαμε να σας βγάλουμε έξω από αυτό. Όχι, εσύ, ούτε ο κύριο Σιρόβικ, η κυρία Ρόμαν από την Κομισιόν. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Ο κύριος Σίμψον ήδη εξήγησε το ιστορικό και πώς καταλήξαμε στην πρόταση αυτή της Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα τώρα να σας εξηγήσω λίγο περισσότερο γιατί από τεχνική σκοπιά θεωρούμε, θεωρούμε τις τελευταίες τροπολογίες από 18 έως 22 δηλαδή γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Οι μεταβλητές αυτές δεν συμφωνούν με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για τον παρόντα κανονισμό. Οι στατιστικές μονάδες στην περίπτωση αυτή αντιπροσωπεύουν στην ουσία τα οχήματα και στις περισσότερες χώρες που κοινοποιούν δεδομένα ο αριθμός οχημάτων είναι μεγάλος. Γι' αυτό και οι κοινοποιούσες χώρες πρέπει να ε, κάνουν μια δειγματοληπτική έρευνα που γίνεται για να συλλεχθούν οι πληροφορίες. Το δείγμα μπορεί να είναι 5 μέχρι 10 το πολύ του συνολικού πληθυσμού και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί το λέω. Γι' αυτό η χώρα μέλος πρέπει να κάνει μια αντιπροσωπευτική επιλογή από τον πληθυσμό αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε και στην βάση των διανυωμένων χιλιόμετρων και μέσα στα πλαίσια μιας ε, ε, αποδεκτής ακρίβειας που σημαίνει βέβαια ότι βασιζόμαστε σε διαφορετικά στάνταρ των στατιστικών θεωριών. Στην πράξη πώς μπορούμε να βρούμε τα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας τις δειγματοληπτικές έρευνες και μετά με ε, ορισμένους σταθμιστικούς παράγοντες οι οποίοι υπολογίζονται σε βάση ορισμένων αρχών και ορισμένοι παράγοντες αυτούς είναι ο τύπος της συλλεγόμενης πληροφορίας και γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος μη συνεπών αποτελεσμάτων. Αν χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αυτούς τους παράγοντες για μεταβλητές οι οποίες δεν βασίζονται στις ίδιες αρχές με αυτές που συλλέγουμε ε, με βάση τον παρόντα κανονισμό. Έχουμε λοιπόν συνολικά δεδομένα στο εθνικό επίπεδο που ενδεχομένως θα είναι μη ακριβή. Να έλθω τώρα στις τροπολογίες 15 έως 17. Η Κομισιόν θεωρεί τις ε, τροπολογίες αυτές καταρχήν αποδεκτές και για τις υπόλοιπες ισχύουν τα σχόλια που σας ανέφερα προηγουμένως. Ο πρόεδρος Σίμψον, σας ευχαριστώ. Τι να προσθέσω εγώ, νομίζω τα είπα όλα. Θα επιμείνω στην αρχική μου θέση. Κύριε Λίχτενμπεργκερ, θέλετε λίγο να λάβετε το λόγο σύντομα. Ναι, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ε, σχετικά με την αντιπαραβολή των διαφόρων στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη. Εάν όμως παραμείνουμε σε μια θέση που θα λέμε που θα λέμε στην ουσία δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δεδομένα, δεν το κάναμε ποτέ έτσι, τότε στην ουσία υποκλεινόμαστε στην διοικητική πρακτική της Αυτοκρατορίας. Καλά, θα ψηφίσουμε αύριο για να δούμε αν θα επιστρέψουμε στην Αυτοκρατορία των Αυσούργων. Σας ευχαριστώ λοιπόν το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη και ευχαριστώ Ρόμπερτ που μπορέσαμε να σας βάλουμε πιο πριν. Θα σας είπαν ότι ο κύριος Κόξ είχε κάποια προβλήματα. Χρειάστηκε λοιπόν να φέρουμε πιο πριν την ε, έκθεσή του και ψάχνουμε να βρούμε μέλη να έρθουν για να συζητήσουμε άλλες εκθέσεις. Χαίρομαι λοιπόν που ήρθατε για τη γνωμοδότησή σας για την εποπτεία της αγοράς για δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας θυμίσω ότι είχαμε κάνει μια πολύ καλή συζήτηση για αυτό το θέμα το Φεβρουάριο και με τον ίδιο θερδικό τρόπο συνεργάστηκα με τους σκιώδεις εισηγητές. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση γενικά για την προσέγγιση στα θέματα που θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή, για τα θέματα δηλαδή οδικής ασφάλειας, για επέκταση του ABS και στα και τις μοτοσικλέτες, ε, να δημιουργήσουμε μια νέα ε, κατηγορία για τις μηχανές ε, enduro και για τις, τις μοτοσικλέτες δοκιμών, να συμπεριλάβουμε και τα οχήματα off crucial point was an extension of mandatory fitting for ABS, uh, and finally, uh, we I think we had a good um, agreement uh, and with the shadows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 Uh, what I can say more on this uh, dossier, I can say uh, there are 13 amendments are tabled after initial draft report, and then we have a. Και τρεις τροπολογίες έχω υποβάλει εγώ, τρεις έχουν υποστηρίξει και άδειες εισηγητές. Οι τρεις είναι του, του κύριου Κράμερ έχουν αποσυρθεί. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, καθώς και τους και για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω ότι νομίζω πως ο κύριος Ζήλ έχει κάνει εξαιρετική έκθεση. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε εδώ και καιρό να κάνουμε, γιατί στην ουσία συγκεντρώνει ε, τέσσερις διαφορετικές οδηγίες. Είναι δηλαδή ένα ε, παγιωμένο κείμενο και πολύ λογικό, όπως είπε και ο εισηγητές κύριος Ζήλε, Θέλουμε λοιπόν να με περιορίσουμε τι εκπομπέ, να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια. Τρίτον, να λάβουμε υπόψη τι νέε τεχνολογίε. Και τέταρτον, να βελτιώσουμε την εποπτεία τη αγορά. Έκανε σπουδαίο έργο, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντίσταση σε αρκετή πίεση από την ίδια τη βιομηχανία, γιατί ένας από τους ε, παράγοντες κόστος που μας τόνισε η βιομηχανία είναι το κόστος του ABS σε αντίθεση με το CBS. Πρόκειται για ένα σύστημα που εμποδίζει το μπλοκάρισμα των φρένων. Εάν δεν έχεις τέτοιο όμως σύστημα, η πιθανότητα ολίσθησης μπορεί να σε φτάσει μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ σοβαρό ατύχημα. Ε, η ασφάλεια είναι λοιπόν το πιο σημαντικό και δεν δεχόμαστε ορισμένες ε, από τις γραμμές που μας έδωσε η βιομηχανία ότι δηλαδή μπορεί να κοστίζει μέχρι και χίλια ευρώ να εγκαταστήσει κανείς ένα σύστημα ABS σε ένα σχετικά φθηνό ε, μοτοσακό. Ε, εγώ όπω γνωρίζω αυτό γίνεται με 100-200 ευρώ maximum. Αλλά άσχετα από το κόστος, ε, ούτως ή άλλως ε, η βιομηχανία θέλει να κερδίζει 70 με 150 ευρώ ανά ε, μοτοσυκλέτα. Η συμβαστική λοιπόν Β νομίζω είναι λογική, την ανέφερε ήδη ο κύριο Ζήλε. Αν τα κάτι μέλη θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο σε κάποια μεταβατική διαδικασία περίοδο θα μπορούσαν να δώσουν μια επιδότηση ώστε να διευκολύνουν τον κόσμο που έχει ε, μοτοσακό να εγκαταστήσει αυτό το σύστημα ABS. Υποστηρίζουμε λοιπόν την έκθεση πλήρως. Έχουμε τρεις τροπολογίες καταθέσει. Τις έχει υποστηρίξει ο κύριος Ζήλε, η κυρία Σέντερ, ο κύριος Στέρξ και εσείς ο ίδιος. Είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι προσαρμόζουμε μια πολύ λογική έκθεση γιατί τέλος στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ο στόχος μας η οδική ασφάλεια, μικρότερη, χαμηλότερες εκπομπές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ όλος ιδιαίτερος τον κύριο Ζήλε για τον διάλογο που έχουμε μεταξύ μας ώστε να ετοιμαστεί η γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής Μεταφορών για τον ε, σχετικό κλάδο, για αυτή την κατηγορία οχημάτων που είναι όλο και περισσότερα σήμερα και συνεχώς αυξάνονται και που χρησιμοποιούν ε, πάρα πολλοί νέοι και όχι μόνο. Υπάρχουν ε, λοιπόν τα οχήματα επίσης παντός εδάφους και γι' αυτό απαιτείται η διευκρίνηση αυτή και για τα οχήματα παντός ε, εδάφους αλλά και για τις μοτοσυκλέτε Enduro και Trial. Πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια. Ε, δείχνουν μεγάλη ευαισθησία οι προτάσεις που έχουμε μπροστά μας για το πώς θα φαίνονται οι μοτοσυκλέτες, πώς προσπαθούν οι κατασκευαστές να φροντίσουν ε, για τα φώτα να ανάβουν πάντα και να υπάρχει αυτόματο σύστημα που σβήνουν. Επίσης, θέλουμε να φροντίσουμε και το σύστημα πέδησης αντιεμπλοκής στο ABS ε, να υπάρχει πάντα σε όλες τις μηχανές. Μην ξεχνάμε ότι είναι οι πιο νέοι που χρησιμοποιούν τέτοιες μοτοσυκλέτες και πρέπει να υπάρχουν όλες οι εγγύσεις για την ασφάλεια. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι θα υπερβάλλουμε στο κόστος, ότι θα επομιστεί τεράστιο κόστος η βιομηχανία κατασκευής των μοτοστικλών αυτών. Κατά τα ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή τον κύριο Σίλε για την κατανόησή του και για τους συμβασμούς που προτείνει. Οι σοσιαλιστές θα στηρίξουν την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος Στέρξ, εκ μέρους του Άλντε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ζήλε για τον τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε πάνω στην έκθεση αυτή. Είναι πάντα δύσκολο όταν υπάρχουν τόσο πολλές διαφορετικές απόψεις πώς θα τις συμβιβάσουμε. Νομίζω όμως ότι καταφέραμε να ιεραρχήσουμε πάρα πολύ καλά τις ανησυχίες μας και το αποτέλεσμα είναι καλό. Θα Είναι πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο, η ασφάλεια στους δρόμους. Από εκεί και πέρα, οι σκιώδες και ο εισηγητής καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είμαστε λογικοί όσον αφορά την βελτίωση της ασφάλειας στους δρόμους, αλλά και την αποσαφήνιση των σχετικών ρυθμίσεων υπέρ της ασφάλειας στους δρόμους. Έγινε μεγάλη συζήτηση για την πέδηση αντιπλοκή στο ΕΜΠΕΣ, αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει στα, σε όλα τα δίκυκλα ή όχι. Νομίζω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποιες καλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Κράμερ, εκ μέρους των Πρασίνων τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Ζήλε, εισηγητή. Ευχαριστώ και για την συνεργασία με τους άλλους σκιώδης Βέβαια η ασφάλεια είναι το κέριο θέμα. Αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη ασφάλεια επιτυγχάνεται εκεί όπου ο κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο τα ποδήλατα. Για παράδειγμα, Δανία και Ολλανδία, όπου οι άνθρωποι κινούνται περισσότερο με ποδήλατα, έχουν τις χαμηλότερες, ε, τα χαμηλότερα νούμερα ατυχημάτων. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, όπου ελάχιστοι χρησιμοποιούν ποδήλατα, έχουν τον υψηλότερο αριθμό νεκρών και τραυματιών στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ελκυστικότερο το ποδήλατο. Υπάρχει και ένα αρνητικό παράδειγμα από την Αυστραλία, όπου είχαν επιβάλει την ε, υποχρέωση να φορά κανείς κράνος και οι άνθρωποι το συνέδεσαν αυτό με κίνδυνο για το ποδήλατο. Και είπαν, α, εφόσον χρειάζεται κάποιος να φορά κράνος, πάει να πει ότι το ποδήλατο είναι επικίνδυνο και το εγκατέλειψαν. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να περάσει ως μήνυμα. Όσο περισσότεροι ποδηλάτες κυκλοφορούν, τόσο ασφαλέστεροι είναι οι δρόμοι. Τώρα, κάτι ακόμα. Οι τροπολογίες μας δηλαδή, τις οποίες αποσύραμε, προέβλεπε η Κομισιόν στην πρότασή της περιορισμό των ηλεκτρικών ποδηλάτων σε 250 βατ και 25 κιλά βάρος και σκεφτήκαμε μήπως δεν είναι απαραίτητα τα κριτήρια αυτά και να μείνουμε μονάχα στην ταχύτητα. Μαζί με τους κοιόδης ηγητές ωστόσο συζητήσαμε και με εκπροσώπους των οργανώσεων ποδηλατών με προσώπους της βιομηχανίας και των ηλεκτρικών ποδηλάτων ότι δεν είναι αυτό το κριτήριο πραγματικά το πλέον σημαντικό αλλά άλλα. Γι' αυτό αποσύρουμε τη δική μας τροπολογία, αφήνουμε την πρόταση της Κομισιόν ως έχει και απευθύνουμε έκκληση στους ενδιαφερόμενους φορείς να εξετάσουν προς τα που ε, κινείται η αγορά αυτή και να επανέλθουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έρχομαι στα όσα είπε ο κύριος Κράμερ. Ο αριθμός χρηστών ε, ηλεκτρικών ποδηλάτων έχει αυξηθεί σημαντικά. Η ασφάλεια αυτών των ηλεκτρικών ποδηλάτων ωστόσο πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. Γι' αυτό θα ήθελα μέτρα ασφάλειας να ληφθούν βεβαίως αλλά να διευκολυνθεί και η πρόσβαση σε τέτοια οχήματα. Όχι μόνο αύξηση της ασφάλειας με λήψη μέτρων αλλά και οι τιμές των ποδηλάτων αυτών να μην είναι υπερβολικά υψηλές. εάν θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός των προσώπων που χρησιμοποιούν τα ποδήλατα αυτά, όπως είπα, πρέπει και η ασφάλειά τους να είναι εγγυημένη, αλλά και η τιμή να μην ε, γίνει υπερβολική λόγω της προσθήκης αυτών των ειδικών συστημάτων παιδίσεως κλπ. Ευχαριστώ. Κομισιόν. Ευχαριστώ Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητές για την εργασία τους. Λίγα σχόλια για τα τρία κύρια θέματα. Πρώτα να ευχαριστήσω για την δύσκολη δουλειά που ε, έγινε για καλύτερη ταξινόμηση των οχημάτων, κυρίως βεβαίως των εκτός ε, δρόμου και σχετικά με τα κριτήρια βέβαια που ασφαλώς και συμβάλλουν σε μια διευκρίνηση του περιεχομένου της οδηγίας και για τώρα αλλά και για το μέλλον για λήψη άλλων μέτρων για τα οχήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τις συσκευές ή χαρακτηριστικά ασφαλείας τονίζουμε ότι συμφωνούμε βέβαια με την αξίωση να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και ιδίως σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια ελαφρών τετράτροχων οχημάτων. Θα το κάνουμε αυτό. Επισημαίνω ωστόσο το εξής. Ως συνολική προσέγγιση θα θέλαμε να συνεχίσει να υπάρχει διάκριση μεταξύ ε, οχημάτων της ελαφράς κατηγορίας λάμδα δηλαδή L και των επιβατικών οχημάτων. Δεν μπορούμε να ισχυριθούμε δηλαδή ότι ένα ελαφρό τετράτροχο έχει, θα έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας με ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Είναι και θέμα δηλαδή μηχανολογικής κατασκευής. Δεν μπορεί να διαθέτει τα ίδια στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή συστημάτων πέδησης που δεν μπλοκάρουν. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια ισορροπία και στη βάση της μελέτης αντικτύπου όπου θεωρούμε ότι η γραμμή που προτείνουμε στην πρότασή μας όντως ανταποκρίνεται, όντως επιτυγχάνει μια θέση ισορροπίας ανάμεσα στα, ε, στις ελαφρές μοτοσυκλέτες και στα σκούτερ γιατί εξετάσαμε και τι αντίκτυπο θα έχει στην τιμή. Γιατί ιδίω για την κίνηση σε αστικά κέντρα υπάρχει σαφώς αυξητική τάση της χρήσης αυτών των οχημάτων και αυτό επηρεάζει την πρότασή μας όταν ε, είπαμε να χρησιμοποιηθούν συστήματα anti-block στις ε, διάφορες οικογένειες εντό εισαγωγικών των οχημάτων τύπου λάμδα. Και σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό και ότι πρέπει με κάθε προσπάθεια να βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίδοση των ελαφρών οχημάτων και ο χρόνος βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο, όπως είδαμε και στις προπαρασκευαστικές μας μελέτες. Αλλά πάλι λόγω και κόστους αλλά και τεχνικής εφαρμοσιμότητας θεωρούμε ότι η πρόταση που κάνουμε για τα ελαφρά και πολύ ελαφρά οχήματα, σκούτερ κλπ. είναι ισορροπημένη. Και ας μην δυσμονούμε ότι για πολύ καιρό τα οχήματα αυτά δεν αναπτύσσονταν με τον ίδιο ταχύ ρυθμό όπως τα επιβατικά αυτοκίνητα για παράδειγμα. Άρα θα χρειαστούν πολλές επενδύσεις, πολλές μελέτες, πολλές τεχνολογικές εξελίξεις και βέβαια χρόνος για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη αυτή. Ευχαριστώ κύριε Ζήλε. για τα συστήματα ABS για τις μοτοσυκλέτες. Όπως θα θυμάστε, είχε γίνει μια αρχική πρόταση δική μου να διακριθούν τα... οι μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται στην κίνηση στα αστικά κέντρα από αυτές που χρησιμοποιούνται εκτός. Έγινε βέβαια εδώ μια συζήτηση και εμείς βέβαια ασφαλώς αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα είναι επίμαχο και ότι δεν έχουν την ίδια άποψη η βιομηχανία και οι καταναλωτές. Αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι ότι πρόκειται, είναι και θέμα ε, προστασίας καταναλωτών και θέλουμε να συνδράμουμε τους ε, συναδέλφους μας ε, της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτού στην προσπάθειά τους. Και βεβαίως ευχαριστώ όλες και όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου για το θέμα αυτό και από τη Γραμματεία. Ευχαριστώ. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρο στην Επιτροπή Μεταφορών. Λίγη εδώ η ημερήσια διάταξη της ε, τακτικής συνεδρίασης. Εάν είναι παρούσες και παρόντες οι συντονιστές, τότε ας αρχίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κύριο Γκρό, και θα επανέλθουμε αύριο σε πλήρη σύνθεση δηλαδή της Επιτροπής για